η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Καλωσορίζω ξανά στο Κοινοβούλιο την κυρία Ζαρίν Χένις Πλάσχαρτ. Καλωσορίσατε. It's Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που σας βλέπω. Πρόεδρε, Επίτροπε, αξιότιμοι βουλευτέ, ε, το 2016 αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη διεθνή κοινότητα για να καταγράψει τα επιτεύγματα του διεθνούς ε, συστήματος ε, επιτήρησης ε, ναρκωτικών και πρόκειται και μια ευκαιρία να δώσουμε μια απάντηση στη, σε μακροπρόθεσμα προβλήματα σε ό,τι αφορά το πλαίσιο των διεθνών ε, συνθήκων. Το ΆΝΓΑΣ, λοιπόν, η έκτακτη συνέντευξη στην Κοινική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να καταρτήσει ένα συγκεκριμένο και στοχευμένο έγγραφο με συγκεκριμένε λειτουργικέ συστάσει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση για να είμαστε πιο ακριβεί. Είμαστε, λοιπόν, υπέρ των εξή προτεραιότητων. Καταρχά, τονίζομαι ότι η ε, συνθήκες του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των ε, ναρκωτικών και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τους ακρογωνιαίους λήθους για το θέμα των ναρκωτικών. Υπάρχει λοιπόν στις διατάξεις της σχετικής συνθήκης ε, επαρκή ευελιξία για να υπάρξει σωστή ανταπόκριση στο θέμα των ναρκωτικών σύμφωνα με τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Κατά δεύτερον, τονίζουμε τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητούμε την κατάργηση της θανατικής ποινή σε ό,τι αφορά εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά ουσιαστικά και την κατάργηση άλλων πρακτικών που δεν συνάδουν με την αρχή τη ε, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, αλληλεγγύη, κράτου δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να τονίζει ότι η θανατική ποινή δεν σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν υπάρχει και αποτρεπτικό παράγοντα για τα ναρκωτικά. Και επίση υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή τη ε, θανατική ποινή για τέτοια ε, εγκλήματα για τα ναρκωτικά δεν πλήρη τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες για το, το σοβαρά εγκλήματα. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε μία προσέγγιση βάσης τεκμηρίων. Χρειάζονται μέτρα προφανώς για τη μείωση και την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μία προσέγγιση βάσης της δημόσιας υγείας, βάση επιστημονικών στοιχείων, με αντικειμενικά συστήματα ε, επιτήρησης και αξιολόγησης οι συνθήκε λοιπόν, οι διεθνεί συνθήκε για τα ναρκωτικά καλούν για μια ισορροπή αντιμετώπιση, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι σε κάποια κράτη τα μέτρα κατά τη ε, εμπορία και τη παραγωγή ε, ε, των ναρκωτικών είναι πιο σημαντικά από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της χρήσης, της κατανάλωσης των ναρκωτικών και της ανάκαμψης της ε, υγείας του ατόμου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δράξουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία που έχουμε να το βελτιώσουμε αυτό. Καλή επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση στα εμπλεκόμενα μέρη να αυξήσουν την ε, πρόσβαση σε μέτρα δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση του HIV και τα μέτρα αυτά έχουν αποδείξει την αξία τους για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Επίσης, θέλουμε εναλλακτική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα μια ολιστικής προσέγγισης για να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της ε, παρανομής τέτοιας ε, φυτών. Επίσης, τονίζουμε τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και της επιστημονικής ε, κοινότητας για τη μείωση των ναρκωτικών. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε την αναγνώριση του ρόλου τη κοινωνία των πολιτών σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ κατά των ναρκωτικών. Αυτέ οι προτεραιότητε αποτυπώνονται στην κοινή θέση του Άγκα του Δεκεμβρίου. Και στο σχετικό έγγραφο η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στενά στις διαπραγματεύσει σε ό,τι αφορά το έγγραφο του τελικό του Άγκα και χαιρόμαστε που το τελικό αυτό έγγραφο περιλαμβάνει ήδη πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δύο σημαντικά ζητήματα ακόμα λείπουν από το έγγραφο αυτό. Καταρχά, μία αναφορά στην καταργήση τη αντική ποινή για τα ναρκωτικά και κατά δεύτερον, έντονη διατύπωση για τα μέτρα μείωση ε, του κινδύνου και των αντικτύπου. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να επιμείνουμε για να συμπεριληφθούν τα δύο αυτά πολύ σημαντικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Υπουργό και τώρα το λόγο έχει η Επιτροπή. Κυρία Μάρμστρομ, σας ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για να πετύχει η ειδική ε, σύνοδος ε, για τα ναρκωτικά του ΟΗΕ και είμαστε πλήρως προσιλωμένοι στην προετοιμασία της. Θα θυμάστε ότι τον Νοέμβριο εγκρίναμε μια κοινή δήλωση μια κοινή θέση για το ε, Άγκος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, πραγματικά είναι χέρι-χέρι με το Συμβούλιο εδώ. Είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ειδική αυτή συνέλευση και θέλει να προωθήσει το παγκόσμια αναγνωρισμένο ο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μείωση ε, της ζήτησης, μείωση της προσφοράς θέλουμε, αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι το ε, εμπόριο στο ίντερνετ ε, ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. Ε, τα είπε και η κυρία Υπουργό, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά. Προτεραιότητα είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατάργηση της θανατικής ποινής για εγκλήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά. Ε, στο διεθνές δίκαιο. Ε, Προτείνουμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανωθεί ε, στο περιθώριο αυτή τη συνόδου μία διάσκεψη για τη θανατική ποινή για να εξηγήσουμε γιατί δεν είναι καλή πολιτική και καλή λύση. Ποτέ δεν είναι καλή η θανατική ποινή, πόσο μάλλον για τα ναρκωτικά. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης αναλογία και αναλογικότητα της ποινική δικαιοσύνης για τους χρήστες ε, ο βασικός ε, στόχος ε, είναι ένα σύστημα που να ελέγχει διεθνώς τα ναρκωτικά. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τη μείωση της ζήτησης, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία, μείωση του κινδύνου, θεραπεία, κοινωνική ένταξη και απεξάρτηση. Είμαστε σε πολύ καλή θέση για να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές και τις εμπειρίες μας υποστηρίξουμε τις συστάσεις ε, που έχουν υποβληθεί. Θέλουμε μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία και συντονισμό για να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε τα εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Ιδιαίτερα τους διακινητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σπάσουν οι δεσμοί ε, μεταξύ του εμπορίου ναρκωτικών, ε, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητε το ξέπλυμα χρήματος. Η Europol συνεισφέρει πάρα πολύ προς το στόχο αυτό, δίνει εμπειρογνώμονες και διευκολύνει την ανταλλαγή πρακτικών και πληροφοριών. Επίσης, ζητούμε αποτελεσματική διεθνή συνεργασία για προκλήσεις όπως είναι ε, το λαθρεμπόριο στο διαδίκτυο και νέες ψυχοτρόπες ουσίες θα πρέπει να βασιζόμαστε σε στοιχεία με έλεγχο και αξιολόγηση αξιόπιστο και τεκμηριωμένων. Έχουμε το αντίστοιχο κέντρο στη Λισαβόνα. Και τέλος, θέλουμε να Θέλουμε να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για τα γυναίκες, για τα παιδιά και για τους νέους. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πρώτη στην υποστήριξη της κοινωνίας ε, των πολιτών σε ό,τι αφορά θέματα εφαρμογής της ε, πολιτικής αυτής. Ε, έχουμε εκπροσώπους από 25 ΜΚΟ και, και μας βοηθούν διαρκώς στη διαδικασία αυτή. Και προσβλέπω λοιπόν στη συζήτηση και θα λάβουμε υπόψη λοιπόν τα σχόλιά σα ε, πολύ προσεκτικά κατά την προετοιμασία τη επόμενη ε, αγκάς. Ευχαριστούμε πολύ λέει Πρόεδρο. και τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση με εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων. Ο κ. Μπόνι για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η διάσκεψη Άγκα θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να προωθηθεί η ευρωπαϊκή προσέγγιση σε σχέση με θέματα ναρκωτικών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της ε, ζήτησης και της ε, προσφοράς και να καταπολεθούμε τα προβλήματα που προκύπτουν από τα ναρκωτικά. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι μοναδική, καθώς ε, καταφέραμε να συντονίσουμε 28 εθνικές αρχές αντιμετώπισης των ναρκωτικών και να ενισχύσουμε τις δράσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για ένα μοντέλο με ειδικό με το ειδικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθηση Ναρκωτικών και Τοξικομανία για την αξιολόγηση του κινδύνου και θα πρέπει να μοιραστούμε τι εμπειρίε μα με τι περιφερειακέ οργανώσει. Ω Ευρώπη, θα πρέπει να προωθήσουμε την κατάργηση τη θανατική ποινή και το δικαίωμα παροχή υγειονομική περίθαλψη στα άτομα που πλήττονται από τα ναρκωτικά. Είναι σημαντικό να αλλάξει η στάση και η νοοτροπία, όχι να στιγματίζεται ο κόσμος που εξαρτάται από τα ναρκωτικά, όχι να τους τιμωρούμε και να τους ε, καθιστούμε υπέτειους, αλλά να είμαστε προληπτικοί στην προσέγγιση μας και να είμαστε ενήμεροι. Τρία σημεία λοιπόν θα ήθελα να τονίσω. Καταρχάς θα πρέπει να αναπτυχθεί μια περαιτέρω ενοποιημένη προσέγγιση με συνεργασία μεταξύ των αρχών για την υγεία, για την δικαιοσύνη και για την, ε, την κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να καταπολεπούμε πιο συντονισμένα το οργανωμένο ε, έγκλημα. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στους νέους τρόπους ε, διανομής ναρκωτικών, λαμβάνοντας υπόψη και το διαδίκτυο, όχι μόνο για τις ε, αρχές επιβολής ε, του νόμου, αλλά και για τους ε, γονείς και για τις οργανώσεις ε, πρόληψης. Και τρίτον, θα πρέπει να κατανοήσουμε το φαινόμενο των νέων ψυχοτρόπων ουσιών, που αποτελούν όλο και μεγαλύτερη απειλή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης και μια δυνατότητα να αντιδρούμε πιο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι πόροι μα, ιδιαίτερα οι πόροι που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθηση Ναρκωτικών και Τοξικομανία θα πρέπει να ενισχυθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το έχω μία μπλε κάρτα από τον κύριο Τζάνι. Την αποδέχεστε. Κύριε Μπόνη, αποτέχεστε παρακαλώ την μπλε κάρτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που δέχεστε την ερώτησή μου. Και συμφωνώ συμφωνώ με τις προπτικές και όλα τα κριτήρια που αναφέρετε, αλλά έχω μία ερώτηση να σας θέσω για ένα ζήτημα και μόνο. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι εναρμονισμένες πολιτικές πραγματικά μπορούν να υποστρεφτούν από εμάς όταν στην Ουγγαρία η πατήτηδα έχει αυξηθεί κατά 50% και τα σχετικά κρούσματα γιατί η κυβέρνηση επιτρέπει προγράμματα αντικατάστασης σε ε, ε, ο κύριος Μπόνι για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις αρμοδιότητες ε, σε θέματα υγείας. Αυτά είναι στα χέρια των κρατών μελών. Πολλές προσπάθειες γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναρμονιστούν, να συντονιστούν κάποιες δράσεις, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Η προώθηση, η συνεργασία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Αλλά, από την άλλη, να έχουμε υπόψη μας ότι πολλά κράτη-μέλη θα καθορίσουν τις δικές του πολιτικές στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σλάιν. Για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην ετήσια έκθεση του 2014, η Εθνική Διεύθυνση κατά της Μαφίας στην Ιταλία θεώρησε ότι έπρεπε να αναγνωρίσει την πλήρη αποτυχία της πολιτικής που άσκησε κατά της χρήσης της ε, κανάβεως, της μαριχουάνας. Και έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες θετικές ε, ενέργειες της απελευθέρωσης ε, κονδυλίων ε, για την απελευθέρωση οικονομικών πόρων για την καταπολέμηση της μαφία κυρίως. Έτσι έχουμε μία συζήτηση πολύ ζωντανή στις θετικές εμπειρίες από χώρες όπως η Ουρουάη όπου μειώθηκαν και τα εγκληματικά φαινόμενα. Αυτό πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ιδιαίτερα εν ώψη της ειδικής συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης των ΟΗΕ, ε, αφιερωμένη στη ε, ναρκωτικά, μια μοναδική ευκαιρία που έχει στο επίκεντρο τους ανθρώπους και την υγεία τους. Ε, να έχουμε το θάρρος να αλλάξουμε πορεία οι πολιτικές καταστολής δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ε, την αγορά την παράνομη, έχουν ε, γεμίσει, πλημμυρίσει τις φυλακές και έχουν ευνοήσει την διακίνηση την παράνομη που έχουν ε, πλουτίσει τους ήδη πολυκατομμυριούχους οι κινητές ναρκωτικών. Ελπίζω πως πια η Ευρώπη θα κάνει τα απαραίτητα βήματα. Ευχαριστώ. Γιούρεκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Δημοσιογεία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που συναποτελούν ε, κοινό αγαθό όλων των εθνών και καμία κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να το παραβεί αυτό και έχει ευθύνη να το προασπίζει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση οργανωσμένου εγκλήματο. Τα άτομα τα οποία εξαρτώνται από τα ναρκωτικά θα πρέπει να βοηθούνται, να λαμβάνουν θεραπεία και όσοι διαπράττουν τα εγκλήματα θα πρέπει να καταπολεμείται. Πραγματικά ως πόλεμος θα πρέπει να ανακηρυχθεί κατά των ατόμων αυτών. Το βασικό μήνυμα που θα πρέπει να δώσουμε στον υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να είναι η κατάργηση της θανατικής ποινής. Αλλά αυτό ακούμε να λένε πολύ. Τι γίνεται όμως με την κατάργηση των στρατιωτικών δυνάμεων στην καταπολέμηση των ε, ναρκωτικών. Τι γίνεται με τους βαρόνους ε, των ναρκωτικών. Ε? Θέλουμε λοιπόν να αποτρέψουμε τις ενέργειες αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σοντεύσκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι. Το θέμα των ναρκωτικών σήμερα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, όπως και το θέμα της ε, μετανάστευσης. Αλλά δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι παραμένει στο υπόβαθρο ακόμα. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στη διεθνή κοινότητα στο διεθνέ προσκήνιο να υπάρχουν και νέε τάσει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αντίδραση και σε διεθνέ επίπεδο. Βλέποντα τα στατιστικά στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι ανακύπτουν καινούργιε μορφέ ναρκωτικών. Το 2014, για παράδειγμα, 101 ναι, εκατομμύρια νέε ουσίε ε, αναφέρθηκαν. Και το φαινόμενο αυτό συνοδεύεται και με αύξηση των εγκληματικών ενεργειών σε ό,τι αφορά την ε, προσφορά ναρκωτικών. Και το πιο επικίνδυνο είναι η παροχή στο διαδίκτυο παράνομων ναρκωτικών. Υπάρχουν χίλια τέτοια καταστήματα ε, στο διαδικτύο στην Ευρώπη όπου ο κόσμος είναι νέοι. Τα παιδιά μπορούν να αγοράσουν ναρκωτικά. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε και ευρωπαϊκές λύσεις αλλά να αναζητήσουμε και παγκόσμιες καθολικές λύσεις και να δράσουμε προληπτικά σε ό,τι αφορά αυτό, μεγάλο αυτό το πρόβλημα. Κύριε Κύρκος, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην, πρώτη, στην προηγούμενη Άγκα, το 1998, αποφασίστηκε για πρώτη φορά η στήριξη και των αστυνομικών μέτρων, αλλά και των μέτρων πρόληψης και θεραπείας. Αυτό όμως δυστυχώς δεν έγινε. Μείναμε στις διακηρύξεις και έτσι φτάσαμε σήμερα το 80% των διαθέσιμων πόρων να διοχετεύεται στις αστυνομικές εκστρατείες, οι οποίες έχουν αποδειχθεί καθολικά αποτυχημένες. Δυστυχώς, το μόνο που προσφέρουν είναι η ψευδέστηση ότι υπάρχει ένας ισχυρός διώκτης, όμως ο βασιλιάς είναι γυμνός. Για να γυρίσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη η προσφορά ε, ε, θεραπείων οι οποίες απευθύνονται σε μικροπαραβάτες χρήστες εναλλακτικές της φυλάκησης. όπως και η προσφορά τέτοιων προγραμμάτων θεραπείας για μέσα στις φυλακές. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσουν τα υποπτευόμενα κέντρα χρήσης, τα οποία όχι μόνο σώζουν ζωές των χρηστών, αλλά εμποδίζουν και τη μετάδοση μολυσματικών νόσων στο γενικό πληθυσμό. Σκεφτείτε, κάθε μία ζωή η οποία σώζεται σε ένα κέντρο υποπτευόμενης χρήσης σημαίνει επιπλέον και ένα ελεύθερο κρεβάτι σε μία μονάδα εντατικής θεραπείας. Ποιο συγγενής ανθρώπου που το έχει ανάγκη δεν θα κλιπαρούσε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ο μιλητής, ο κύριος Πόλτσακ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τον προηγούμενο μελητή σε ό,τι αφορά το ρόλο της πρόληψης και του μη αποκλεισμού των ανθρώπων που εξαρτώνται από τα ναρκωτικά και ε, εκ παραλλήλου υπάρχουν και οι οργανώσεις ε, που θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν για να επανενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι στην ε, φυσιολογική κανονική ζωή. Σε παράλληλα, θα ήθελα να σας υπογραμμίσω και το θέμα του ποινικού δικαίου, γιατί εδώ έχουμε και προβλήματα των καινούριων ουσιών που παρέχονται και οι οποίες ε, μάλιστα εντοπίζονται και στον ευρωπαϊκό χώρο. Το τελευταίο έτος ε, ήταν 23 τόνοι αυτοί λοιπόν που εντοπίστηκαν. Μιλάμε για τεράστιους, τεράστιες ποσότητες. Θα πρέπει λοιπόν να εντοπίζονται, να περιγράφονται οι ουσίες αυτές και το θέμα είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, προσφορά των ουσιών αυτών. Ποια είναι λοιπόν η εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην διασκέψη του ΟΗΕ και Ποια θέση θα εκπροσωπήσουμε. Ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη λοιπόν και αυτά τα νέα, αυτές οι νέες ουσίες Τώρα λοιπόν στη διαδικασία Καρσδεάη ο κύριο Καπούτο πρώτος. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχει μια πτυχή που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη από τη ε, στρατηγική ε, καταπολέμηση των ε, ναρκωτικών. Δεν είναι οι δυνατότητε καταστολή, αλλά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ναρκωτικών το 2015 εκατομμύρια εκτάρια καταστράφηκαν στη Λατινική Αμερική για να καλλιεργηθεί η κοκαίνη. Σύμφωνα με διάφορες ΜΚΟ, στις πιο κρίσιμες περιοχές, οι περιβαλλοντικές ε, επιπτώσεις ε, της καλλιέργειας των ναρκωτικών είναι πιο σημαντικές από ότι αυτές των κλιματικών αλλαγών. Θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική εναλλακτική επιλογή για τους ε, καλλιεργητές ε, ναρκωτικών. Γι' αυτό και θα πρέπει να σκεφτούμε αυτό το θέμα, το οποίο θίγεται από ανεξάρτητες μελέτες διαφόρων οργανισμών. Μόνο έτσι θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε όλες τις πτυχές των ναρκωτικών και όχι μόνο το θέμα της καταστολής. Ευχαριστώ. Κύριος Μαριάς κυρία πρόεδρε σε μια φάση τεράστιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης φτώχειας και ανεργίας σε μια φάση έντασης των παγκόσμιων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών σε μια φάση επιδείνωσης της κοινωνικής συνοχής της μεγαλοπόλης της ευρώπης των ΗΠΑ τη της ασίας και της λατινικής αμερικής σε μια φάση ενίσχυσης του λαθρεμπορίου της εγκληματικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών η συνδιάσκεψη του οηε για τα ναρκωτικά θα μπορούσε υπό όρους και προϋποθέσεις να αποτελέσει μια ελπιδοφόρα ακτίδα φωτός μια ευκαιρία για παγκόσμια συνεργασία πρώτον στο χτύπημα του εμπορίου αλλά και της καλλιέργειας ναρκωτικών δεύτερον στην επιβολή σκληρών ποινών και μηδενικής ανοχής στους εμπόρους ναρκωτικών τρίτον στο χτύπημα των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών on the spot αλλά και στο διαδίκτυο τέταρτο στη διαμόρφωση μιας πολιτικής που θα συμβάλλει στην πρόληψη και στην ενημέρωση της νεολαίας για τη μάστιγα των ναρκωτικών και πέμπτον στην ενίσχυση διαδικασιών απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης. Οψόμεθα λοιπόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάκοφτσης Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, είναι καλό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με 28 σαφείς ψήφους υπέρ ενέκρινε ε, και θα ε, παρακολουθήσει αυτή την έκτακτη διάσκεψη του ΟΗΕ. Έχουμε ε, εμπειρία σε αυτά τα θέματα, στην επανένταξη, στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, Έχουμε το ρόλο ε, των συστημάτων υγείας. Έχουμε διάφορες εκστρατείες σε πολλές περιφέρειες και σε πολλές πόλεις ε, κατά πολέμηση των ναρκωτικών. Ξέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά πράγματα για τα ναρκωτικά και ε, μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις εμπειρίες με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης και η Ευρωπόλ έχει τις δικές της εμπειρίες και μπορεί να βοηθήσει. Βέβαια πάντα θα πρέπει να επιλέγουμε την πρόληψη όταν καλούμεθα να αποφασίσουμε και να επιλέξουμε μεταξύ πρόληψης και καταστόλης. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ ευρύ η ατζέντα που θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο αυτό στην Νέα ε, Υόρκη την Άνοιξη, τα πιο πολλά από τα θέματα τα οποία θίξατε, περιλαμβάνοντας την ημερήσια διαταξή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα θέσει σε ό,τι αφορά την πώληση ε, online, τις νέες πολιτικές, νομίζω ότι ε, εντοπίζεται από το Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών ε, μια νέα ουσία κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, τα θέματα της πρόβλεψης, τα θέματα της αντιμετώπιση τη περίθαλψη κτλ. Η αξιότιμη βουλευτή ε, από την Ιταλία μίλησε για την αποποινικοποίηση. Διάφορε χώρες, ξέρετε, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Το θέμα αυτό δεν έχει μπει στην ατζέντα, αλλά ασφαλώ και θα ακούσουμε τις διαφορετικές ε, ε, απόψει των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο. Πολλά λοιπόν έχουμε να συζητήσουμε και θα εξασφαλίσω, θα, θα φροντίσω να συνεχίσει να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην διαδικασία αυτή σε ό,τι αφορά και την... το μήνυμα αυτό θα το διαβιβάσω στον Επιτρόπο Αβραμόπουλο που θα μας εκπροσωπήσει εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργά να συμβάλλει στην συνεδρίαση Άγκα προκειμένου να προωθήσουμε τις παγκόσμιες λύσεις σε αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την πολιτική διακήρυξη του ΟΗΕ που προ βλέπετε για το 2019. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, Madam Chair. Um... Υπουργός, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπε η κυρία Επίτροπος, Περισσότερα από τα θέματα που αναφερθήκατε, τα περισσότερα από αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη. Βεβαίως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βεβαιωθούμε ότι η Άγκας θα ακολουθήσει το δρόμο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχουμε ε, μια προσέγγιση βασιζόμενη στην υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα ναρκωτικά. Ε, επίσης, διατρανώνουμε και την αντίθεσή μας με τη θανατική ποινή για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και λέμε ότι ούτε αναλογική είναι ούτε αποτελεσματική η θανατική ποινή για τέτοια κακουργήματα. Ε, θα πρέπει να είναι και η διατύπωση πάρα πολύ στεναρή. Έχουμε αποδείξει ότι τα μέτρα που έχουμε εμείς λειτουργούν και αποδίδουν και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τα χρησιμοποιήσουμε και καμία δικαιολογία να δεν τα χρησιμοποιήσουμε για την προστασία της υγείας των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Και εγώ σε αυτό ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Καλή σας τύχη εκεί. Λήξη της συζήτηση αυτής και πάμε στο επόμενο.